βραβεύσει την Εστονία και να δείξει ότι μπορούμε να αναζωογονήσουμε την Ευρωζώνη. Κλείνει η συζήτηση και η ψηφοφορία θα γίνει την Τετάρτη. Και τώρα πάμε στο επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξης. Στις παρεμβάσεις διάρκειας ενός λεπτού, με βάση το άρθρο 150, ο πρώτος στο κατάλογό μου είναι η κυρία Αντωνέσκου. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Στη Ρουμανία, όπως και σε πολλά άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν τα λεγόμενα dream shops ε, τα οποία πολλούν ως υποκατάστατα φαρμάκων κάποιες άλλες ε, κάποιες ουσίες. Υπάρχουν κάποιες, ε, κάποιοι κανονισμοί στη Ρουμανία για την απαγόρευση των ουσιών αυτών. Λόγω όμως της λειτουργίας αυτών των, φαρμα, αυτών των καταστημάτων έχουμε ακόμη την απειλή των ουσιών αυτών και πουσία γενικών αντιδράσεων από τα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είχαμε ε, τις κατάλληλες εξελίξεις. Υπάρχουν λοιπόν ε, άτομα που κινδυνεύουν από αυτές τις ουσίες. Ε, υπάρχουν πραγματικά πολλές χημικώς ε, ε κτηθείς ουσίες. Θα πρέπει να απαγορευτούν. Όχι μέσω της σταδιακής απαγόρευσης. Αυτό δεν είναι λύση. Εμείς θεωρούμε ότι ε, το φαινόμενο αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Δεν θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε όταν θα είναι πλέον αργά. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουν ε, την πρωτοβουλία ε, τα θεσμικά όργανα να καταπολεμήσουν αυτά τα, τα ναρκωτικά αλλά και τα υποκατάστατά τους. Μικρόφωνο. Τώρα, μ' ακούτε. Ευχαριστώ πρόεδρε. Στη Ρουμανία συνεχίζουμε να συνεχίζει η κυβέρνηση, η δεξιά κυβέρνηση να παίρνει κατασταλτικά μέσα μέτρα. Πλήττεται η ελευθερία έκφραση. Στην Ρουμανία η λειτουργία της, της κρατικής τηλεόρασης είναι απαράδεκτη. Ε, το σχέδιο νόμου στην ε, Ρουμανία απαγορεύει το δικαίωμα της έκφρασης των μειονοτήτων και αντιβαίνει στο Σύνταγμα. Η αντιπολίτευση κατήγγειλε την ε, πολιτική αυτή και το γεγονός ότι έρχεται σε αντίθεση με το άρθρο 10 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων των, των Ανθρώπων. Ζητώ από τις ε, ρουμανικές αρχές να βρουν ένα μηχανισμό που θα επιτρέψει στην δημόσια ραδιοτηλεόραση να λειτουργήσει βάσει των ευρωπαϊκών αρχών. Κύριε Αλφάνο. Μισό λεπτό, Πρόεδρε. Questo è quello che accadrebbe se in Italia una legge presentata αυτό θα συνέβαινε αν ε, στην Ιταλία ένας νόμος που, ε, ναι, που ενέκρινε η γερουσία την περασμένη εβδομάδα περάσει και στο, στη Βουλή. Με τον νόμο αυτό, οποιοδήποτε δημοσιεύσει ε, υποκλοπές τηλεφωνικές καταδικάζεται. Αυτό είναι αντισυνταγματικό και αντιβαίνει στην ΕΣΔΑ. Το άρθρο 11 της ΕΣΔΑ προβλέπει ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα ελευθερίας έκφρασης και να ενημερώνεται και να παίρνει πληροφορίε. Εγώ ένα παράδειγμα θέλω να σα δώσω μόνο, ε, γιατί είναι πραγματικά μια μορφή ε, λογοκρισίας με ένα παράδειγμα. Ο πατέρα μου ήταν δημοσιογράφος, δολοφονήθηκε από τη μαφία. Τα τελευταία 7 χρόνια, χάρη στι υποκλοπε, διαπιστώθηκε ποιο είχε δώσει την εντολή αυτή τη δολοφονία. Χάρη στην παρακολούθηση αυτή των υποκλοπών, ε, μάθαμε γιατί σκοτώθηκε ο άνθρωπος αυτός. Παρακαλώ τα ευρωπαϊκά όργανα να προσέξουν την κατάσταση. Ο κύριος Νίκολσον. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να επισημάνω την κρίση που αντιμετωπίζουμε στην τοπική κυβέρνηση της Βόρειας Ιρλανδίας όπου είχαμε ένα πρόστιμο άνω των 60 εκατομμυρίων ευρώ για τα λεγόμενες επιδοτήσεις σε στις ε, ενιαίες πληρωμές ε, σε αγρότες. Βεβαίως, λαμβάνω πως πρέπει να τηρούμε τους κανόνες. Να πω εδώ πέρα πως ε, τα χρήματα τα οποία είχαν καταβληθεί αχρεωστητός ήταν 3 εκατομμύρια σε διάρκεια 5 ετών. Οπότε πρόκειται για μια απόφαση άδικη και βεβαίως επιβάλλει ένα πρόστιμο καταποκοπήν και όχι αναλογικό. Γνωρίζουμε ναι. όλοι βεβαίω τα προβλήματα που έχουν οι κυβερνήσει με του προπολογισμού σε όλη την Ευρώπη και οπωσδήποτε τα δημόσια οικονομικά τη Βόρειας Ιρλανδία θα υποφέρουν. Τώρα δεν ξέρω ποιο φταίει κυρία Πρόεδρε, αλλά ξέρω πω οπωσδήποτε δεν φταίνε οι αγρότε. Αλλά αυτό ο οποίο θα πληρώσει είναι ο προπολογισμό τη Βορειοϊρλανδίας σε εποχέ δύσκολε. Ευχαριστώ κύριο Σόντεργαρτ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο Μπούζεκ για το ότι ανέφερε στην εισαγωγή του την κατάσταση στο Ιράν και το ότι είναι ανησυχητική. Οπωσδήποτε ήταν και διπλωματικός. Η κατάσταση εκεί πέρα είναι καταστροφική. Οι αγωνιστές της δημοκρατίας φυλακίζονται, συνδικαλιστές φυλακίζονται, άλλοι άνθρωποι ρίχνονται στη φυλακή με παράλογες κατηγορίες και μένουν εκεί πέρα χρόνια και κάθε μέρα έχουμε νέες καταδίκες. για να καταπιεστεί οποιαδήποτε κριτική της αντιπολίτευσης όλα αυτά. Από την τελευταία μας δε ολομέλεια είχαμε την ε, επίσκεψη ενός ε, Υπουργού και θα ήθελα να γνωρίζω ποια είναι η άποψη του Προεδρείου. Ο κύριος Βαντίμ Τουντόρ. Πρόεδρε, πριν από λίγες εβδομάδες ε, η πρώην ε, νύφη της βασίλισσας της Βρετανίας, η δούξα της ε, πέρασε στα πρωτοσέλιδα γιατί δήλωσε 500.000, ε, ζήτησε 500.000 σελίδες για να, πληροφο, για να δώσει πρόσβαση στον πρώην σύζυγό της, τον πρίγκιπα Ανδρέα. Η συγνώμη που έδωσε μετά δεν, απο, δεν μας αλλάζει την άποψη. Αυτό είναι πολύ κοινό πολύ σύνηθες και γίνεται πάντα. Η, δείχνει πόσο τεχνο, το τεχνολογικό θαύμα των κρυμμένων των κρυφών καμερών. Μια χώρα που δεν θα έβλεπε ποτέ αυτά τα πράγματα τώρα μπορεί να τα δει. Πριν από 200 χρόνια ο Ναπολέων πήρε ένα ε, έγραψε στο, στη Διαθήκη του στην Αγία Ελένη ότι του αφήνει ένα ασημένιο ρολόι σαν ε, ανάμνηση από τον πόλεμο. Αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί τώρα ως ε, διαφθορά. Ευχαριστώ πρόεδρε. Με την ευκαιρία του λεπτού θα ήθελα να συγχαρώ την Ισπανική Προεδρία για τις προσπάθειες που κατέβαλε κατά το εξάμεινο αυτό για να ξεπεραστεί η κοινή θέση σε σχέση με την Κούβα και να δημιουργηθούν νέες σχέσεις μεταξύ Ένωσης και Κούβας που θα περιλαμβάνει βέβαια ως ε, βασική προτεραιότητα την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Η πολιτική αυτή δεν στέφθηκε από επιτυχία κυρίως λόγω της ε, αδιαλαξίας της κουβανικής δικτατορίας. Η Προεδρία ξεκίνησε τον Ιανουάριο με την απέλαση του υποφαινόμενου όταν ε, ε, θέλησαμε να επισκεφθώ, θέλησα να επισκεφθώ νομιμότατα και με θεώρηση στο νησί για να ασχοληθώ με τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκεί. Η νέα αυτή πολιτική ωστόσο που ξεκίνησε η Ισπανική κυβέρνηση θα δώσει ε, αργά ή γρήγορα αποτελέσματα. Ευχαριστώ. κύριος Κόσλικ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε η νέα δεξιά κυβέρνηση της Ουγγαρίας ε, του κυρίου Όρμπαν που έχει πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο ακολουθεί μια εθνικιστική πολιτική. Πρώτος νόμος που έφερε στο Κοινοβούλιο αφορούσε την διπλή υπηκότητα που δίνει την δυνατότητα σε ανθρώπους Ούγγρους ε, το γένος να αποκτήσουν ε, σε άλλες χώρες να αποκτήσουν ε, ουγγρικό διαβατήριο. Ε, μιλάμε δηλαδή για εξοδαφικότητα και αρνείται και να το συζητήσει με τις γειτονικές χώρες η Ουγγαρία. Παραβιάζεται λοιπόν κάθε αρχή της συνύπαρξης των ε, εθνών και εδώ πέρα πλέον αμφισβητείται η συνθήκη του Τρίανου και είναι ένα προειδοποιητικό σημάδι για την Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ο κύριος Χουντής. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Βάσει των πληροφοριών από τον Ιταλικό τύπο, στις 31 Μαΐου, μια Ιταλική ασφαλιστική ε, εταιρεία ε, επέβαλε έναν εθνικό, μια εθνική ε, επιδότηση αυξάνοντας, υποχρεώνοντας μάλλον βούλγαρους πολίτες να πληρώσουν μεγαλύτερα ασφάλιστρα. Ε, η εθνική πολιτική Ωστόσο και η ευρωπαϊκή πολιτική ε, απαιτεί ισότιμη μεταχείριση των ε, ασφαλιζομένων εξάρτητα από την εθνική τους καταγωγή. Είναι μια τέτοια πρακτική σύμφωνη με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία κατά των διακρίσεων. Ευχαριστώ κυρία Γιώτοβα. Πρόεδρε, θα μιλούσα για το Σέγγεν. Άλλο πράγμα θα σας πω όμως. δίνεται εξουσία στην Eurostat για να εξεταστούν, για να παρακολουθούν το, τον προπολογισμό της Ένωσης. Όλοι η ΡΕΝ θα στείλει στη Βουλγαρία την πρώτη ελεκτική επιτροπή του για να εξετάσει την ευθύνη ε, των βουλγαρικών στατιστικών δεδομένων στο δημοσιονομικό έλλειμμα της χώρας σε δύο μέρες η θέση της Βουλγαρίας στις διεθνείς αγορές δινώθηκε φοβερά. Εμείς υποστηρίζουμε τις νέες εξουσίες της Eurostat. Πιστεύουμε ωστόσο ότι θα έπρεπε να, δεν θα έπρεπε να παρουσιάζονται προκαταρκτικές απόψεις για μια χώρα που ενδεχομένα να βλάψουν την εικόνα της προς τα έξω. Πρέπει πρώτα πρώτα να υπάρχει μια ανάλυση για το αν υπήρξε κατάχρηση ή όχι. Προφανώς η βευγανική βεβουλγανικη κυβερνηση δεν είχε σωστή επικοινωνιακή πολιτική με την ε, Κομισιόν. Δεν είναι σωστό ωστόσο να χρησιμοποιούνται οι χώρες για να ενισχύεται η δυνατότητα της Ένωσης να αποκτήσει περισσότερες εξουσίες. Κυρία Παρβάνοβα. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, οι διαμαρτυρίες που ακολούθησαν τις προεδρικές εκλογές ε, του Ιουνίου 2009 αποτέλεσαν αφορμή έτσι ώστε το καθεστώς να συνεχίσει να παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των γενικών σύμφωνα πολλές οργανώσει και την Διεθνή Αμνηστία. Ο αρχηγός του κράτους, η επαναστατική φρουρά και άλλες ε, αρχές συνέχισαν την πρακτική των προηγουμένων ετών. Παρά την απελευθέρωση 89 κρατουμένων φημολογείται πως 450 άλλοι κρατούμενοι παραμένουν στις φυλακές μετά από τις δίκες που ακολούθησαν τις εκλογές. Είχαμε δε τον Ιούνιο μόνο 22 εκτελέσεις. Πρέπει να στείλουμε λοιπόν ένα ισχυρό μήνυμα αλληλεγγύη στον Ιρανικό λαό. Δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια στις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και σύμφωνα με το ψήφισμα της 10 του 2010 πρέπει να δώσουμε προσωρινό άσυλο στους ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θα πρέπει να ζητήσει αναστολή της θανατικής ποινή σύμφωνα με τις αποφάσεις του. Ευχαριστώ κυρία Ντότζ. Uh, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να διατυπώσω την ανησυχία μου για τα αυξανόμενα επίπεδα τρομοκρατία στη Βόρεια Ιρλανδία πρόσφατα. Ορισμένοι από εσά ίσω γνωρίζετε την πρόσφατη δολοφονία του Μπόμπι Μόφατ. Τον δολοφόνησαν αυτοί οι οποίοι, υποτίθεται ότι σχετίζονται με παραστρατικούς το μεσημέρι στο Μπελφάστ όταν οι κανονικοί άνθρωποι πηγαίνανε στις δουλειές τους. Πιστεύουν αυτοί, λίγοι μεν, ότι μπορούν ε, με αυτόν τον τρόπο να ε, επιβάλλουν δικαιοσύνη. Ένας αστυνόμος της Βόρειας Ιρλανδίας είπε ότι η απειλή από την τρομοκρατία στη Βόρεια Ιρλανδία είναι στα χειρότερα επίπεδα εδώ και χρόνια. Ελπίζω ότι οι κοινοβουλευτικοί οι βουλευτές θα συμφωνήσουν ότι τάσσονται στην πλευρά των καλών ανθρώπων της Shackle Road και των της πλειοψηφίας των Ιρλανδών ε, που έχουν αγανακτήσει με αυτή τη δολοφονία και είναι αντίθετη με τροποκρατία. Ο κύριος Τεξέρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μία συμφωνία ελευθερίου, ελευθέρου εμπορίου συνήφθηκε με τη, μεταξύ Κολομβίας και καλύπτοντας βασικά αγροτικά προϊόντα, μπανάνες, ζάχαρη, ε, που είναι πολύ σημαντικά προϊόντα για τις υπερ απομακρυσμένες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτές οι περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, ε, πολύ απομακρυσμένε είναι πολύ Οι Οι Κανάριοι νήσοι χάσανε ένα 20% της αγοράς Μπανάνα πρόσφατα. Θα θέλαμε λοιπόν να γίνει σωστή αξιολόγηση τη συμφωνίας ώστε να ξέρουμε τι επιπτώσεις έχει αυτή η συμφωνία παραδείγματο χάρη στις Καναρίους νήσου. Θα θέλαμε κάποια αντισταθμιστικά μέτρα. Η κυρία Μπάουερ τώρα. Κυρία... Πρόεδρε, η Κεντρική Ευρώπη υποφέρει από τις πλημμύρες. Η Ουγγαρία, Σλοβακία και Τσεχία έζησαν μεγάλες καταστροφές. Γι' αυτό απαιτείται η αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης το συντομότερο δυνατό. Πρέπει λοιπόν να καταβάλει κάθε προσπάθεια η Ένωση για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις ζημιές. Κανένα κράτος μέλος δεν μπορεί να το κάνει αυτό μόνο του. Το δεύτερο πρόβλημα το οποίο θα ήθελα να αναφέρω είναι η διάκριση λόγω του νόμου περί υπηκότητας της Σλοβακίας. Σύμφωνα με το νέο νόμο, όσοι έχουν διπλή υπηκότητα από 17 Ιουλίου δεν θα έχουν πρόσβαση πλέον σε κάποιες θέσεις εργασίας ανεξαρτήτως του από ποια χώρα προέρχονται. Και παραδείγματος χάρη δεν θα μπορέσουν πλέον να έχουν πρόσβαση ε, στις δημόσιες υπηρεσίες, να γίνουν δημόσιοι υπάλληλοι και βέβαια αυτό αποτελεί κίνδυνο για το κράτος ε, και είναι απολύτως απαράδεκτο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Τικάου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. η Κομισιόν και τα κράτη-μέλη πρέπει να επεξετάσουν το, το, τα, τα καινούργια, να αναθεωρήσουν τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών, διότι αυτά αποτελούν σημαντικό κομμάτι της Στρατηγικής Ένωσης για το 2020 και την κοινωνική και οικονομική συνοχή της Ένωσης. Πρέπει να υπάρχουν δίκτυα αποτελεσματικά και πραγματικά λειτουργικά με σιδηρόδρομους υψηλής ταχύτητας που θα επιτρέπουν τη μετακίνηση όλων των Ευρωπαίων ε, πολιτών και την, τον εξυγχρονισμό ταυτόχρονα λιμένων τόσο στη θάλασσα όσο και στα ποτάμια. Ταυτόχρονα θα πρέπει να επανεξεταστούν τα κονδύλια για την ε, να αυξηθούν τα κονδύλια τα σχετικά από το 11% του συνόλου των πολιτικών συνοχής στο 20% ιδίως δε στην κεντρική και νότια Ευρώπη. Θα πρέπει να δοθεί έμφαση στις επενδύσεις ε, στα κράτη-μέλη με απέτηση αύξησης της χρηματοδότησης από την Ένωση. Ευχαριστώ κύριος Βότσον. Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να επισύρω την προσοχή στον αποκλεισμό στο Μανιπούρ, στην Ινδία. Ο αυτοκινητόδρομος 39 έχει μπλοκαριστεί από τις 20 Απριλίου και δεν υπάρχουν μεταφορές φαρμακευτικών ειδών και πετρελαίου και ενέργειας για όλο τον πληθυσμό. Τα νοσοκομεία μπορούν να αντιμετωπίσουν μόνο τα καταπήγοντα και οι τιμές ανέβηκαν κατά 300% στη μαύρη αγορά και μισό εκατομμύριο παιδιά είναι τα, αυτά τα οποία υφίστανται τη μεγαλύτερη βλάμα. βλάβη. Με Πρόκειται για φιλή νάγκα και φοιτητέ νάγκα που έχουν αποκλείσει αυτόν τον αυτοκινητόδρομο. Ελπίζω να με βοηθήσετε ώστε να ζητήσουμε από την ειδική κυβέρνηση να ζητήσουμε διευθέτηση και απόσυρση των ειδικών εξουσιών των στρατιωτικών δυνάμεων ώστε να σταματήσει η ανθρωπιστική κρίση που είναι τόσο σημαντική όσο και στη Γάζα θα έλεγα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τόλκες. Κυρία Πρόεδρε, σε ό,τι φορά την Ουγγαρία και την Σλοβακία, οι χώρες αυτές αντιμετωπίζουν πλημμύρες, τεράστιες πλημμύρες και στις δύο χώρες ωστόσο υπήρξαν, είχαμε κοινοβουλευτικές εκλογές. Αυτό μου θυμίζει μια μεταφορά. Πρέπει να βοηθήσουμε την περιοχή με συντονισμό των δράσεων. Σε ό,τι αφορά τις δύο αυτές χώρε, δεν αφο... δεν... η σκέψη μα δεν πρέπει να αφορά μόνο τη Σλοβακία και την Ουγγαρία, αλλά όλες τις χώρε της κεντρική ε, ε, Ευρώπης και τη Ρουμανία που περνάει ακόμα μια μετακομμουνιστική κρίση. Πρέπει να σας πω ότι πάντα σκέφτομαι τα θύματα της, ε, των πλημμυρών και ζητώ το Κοινοβούλιο να, υποστη, να υποστηρίξει ταχεία βοήθεια σε αυτού. Σε ό,τι αφορά τις εκλογές, χαίρο διότι μαθαίνω, το, διαπιστώνω τα αποτελέσματα, τα αντικομουνιστικά αποτελέσματα. Ζητώ από το Κοινοβούλιο να μας βοηθήσει στη μάχη κατά της ε, κομμουνιστικής κληρονομιάς που δημιουργεί τις κρίσεις. Ευχαριστώ. κύριος Κίτας, ευχαριστώ. Η Κομισιόν προετοιμάζει μία πράσινη βίβλο για τις συντάξεις για να ξεκινήσει μία συζήτηση και θα προσπαθήσει να λύσει το δημογραφικό πρόβλημα και το δημοσιονομικό πρόβλημα των κρατών μελών. Δεδομένου το ότι έχουμε έναν πληθυσμό ο οποίος γυράσκει βεβαίως θα συνεχίσουν να υπάρχουν πιέσεις και ανεξαρτήτως των πολιτικών πιέσεων θα πρέπει να εγγυηθούμε αξιοπρεπή διαβίωση για τους συνταξιούχους. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως είναι μια ομάδα που δεν μπορεί να αμυνθεί και δεν έχουν άλλη πηγή εισοδήματος λόγω της ηλικίας τους, οπότε θα επιμείνω αυτή να είναι η πρώτη προτεραιότητα αυτού του εγγράφου. Κύριος Ματσάρος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μιλάμε αυτές τις μέρες για την ειρήνη του Τριανών, τη συνθήκη του Τριανών που συμπλήρωσε 90 χρόνια. Όταν ε, μετά την υπογραφή της συνθήκης του Τρενών, χιλιάδες, εκατομμύρια Ούγγρων βρέθηκαν σε ξένες χώρες. Η χώρα μας έχασε τα δύο τρίτα του εδάφους της. Αυτό είναι άδικο, όντως. Ωστόσο, πρέπει να δεχθούμε με τα ταπνοφροσύνη την κατάσταση. Δεν θέλουμε να αλλάξουμε τα σύνορα προφανώς. Απλά ζητάμε να υπάρξει σεβασμός της γλώσσες και του πολιτισμού μας εμείς οι Ούγγροι που ζούμε στην Σλοβακία δεν είμαστε ικανοποιημένοι από την κατάσταση. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη γλώσσα μας. Σε ό,τι αφορά δε την απόφαση της Ουγγαρίας για τη διπλή ηθαγένεια, πρόκειται για κάτι συμβολικό για μας. Σημαίνει κάτι για όλους τους Ούγγρους, δεν, έχει, δεν συνιστά καμία απειλή για άλλες χώρες. Θα ήθελα να ζητήσω λοιπόν από τη Σλοβακία να καταστήσει δυνατή την χορήγηση της διπλής ηθαγένειας. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να μιλήσω για την καταπολέμηση της φτώχειας σε αυτό το ευρωπαϊκό έτος. Κατά την συνδιάσκεψη των Υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικών Υπηρεσιών μιλάμε για, μιλήσανε για 20 εκατομμύρια ανθρώπους που είναι σε κατάσταση φτώχειας. Αυτό επικυρώθηκε από τους Υπουργούς. αυτό το θέμα ήταν από τους βασικούς στόχους της Ρέτα Φόλιν Αντιπροέδρου της Κομισιόν και έχω υποστηρίξει αυτή την τοποθέτηση και στο Ευρωκοινοβούλιο κυρία Καλίνξ συνέχισε τις προσπάθειές της η βελγική κυβέρνηση θέλει να καταφέρει να προχωρήσει θετικά την προεδρία της παρά τα θεσμικά μας προβλήματα. Με βάση τα εκλογικά μας αποτελέσματα, η μελλοντική Προεδρία του Βελγίου θα είναι δραστήρια για την υλοποίηση των κοινωνικών στόχων. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λούεν τώρα. Ε, ε. Πάλι είχαμε πλημμύρες στο Δούναβι. Πάλι είχαμε καταστροφές. Η κατάσταση πρέπει να αντιμετωπιστεί και να εξεταστεί από την στρατηγική της Ένωσης για το Δούναβι. Στη συζητήσεις και στην Κωνσταντσα τονίστηκε η ανάγκη τα κράτη-μέλη να δίνουν έμφαση στην οικονομική και κοινωνική διάσταση της λεκάνης του Δουναβού. Οι προτάσεις αυτές θα πρέπει να συνεχιστούν με καινοτόμα μέτρα για να μειωθούν οι ζημιές που προκάλεσαν οι πλημμύρες. Η δεμή, η περιοχή θα αντιμετωπίζει όλο ένα και περισσότερες ζημιές λόγω της μείωσης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και της μείωσης της αναπτυξιακής δυνατότητας. Οι περιοχές αυτές χρειάζονται την ευρωπαϊκή υποστήριξη για να καλύψουν τις ε, ζημιές και να ελαχιστοποιήσουν την καταστροφή. Ο κύριος Σικλούνα. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να μιλήσω για στο Κοινοβούλιο για ένα σημαντικό θέμα το οποίο αφορά τα δημοκρατικά δικαιώματα και την ελευθερία του λόγου. Είναι η ευθύνη μου να εφαρμόζω τα δημοκρατικά μου δικαιώματα και να ενημερώνω τους πολίτες για τις προσπάθειές μου μέσω των media ο ρυθμιστής των μίντια πρέπει να εξασφαλίζει ισορροπία μεταξύ των ιδιωτικών καναλιών γενικά και των μέσων ενημέρωσης. Δεν ζητά βεβαίως ισορροπία για κάθε πρόγραμμα. Δεν σημαίνει αυτό ότι δεν μπορεί κανείς να λάβει το λόγο και να πει τις απόψεις του. Παρόλα αυτά, τρεις φορές με έχουν καταγγείλει ότι έχω παραβιάσει τον νόμο, τον νόμο και γίνεται λογοκρισία των προσπαθειών μου στο Ευρωκοινοβούλιο. Παρόλα αυτά, ε, η ισορροπία δεν αναζητείται μέσω του πλουραλισμού πρέπει να σας πω και της ενθάρρυνσης των διαφόρων πολιτικών απόψεων να διατυπωθούν. Η προσπάθεια είναι να σοπάσουν, να σιγάσουν αυτοί που θέλουν να εκφραστούν. Πολλοί είχαμε μεγάλες φιλοδοξίες όσον αφορά την ένταξη της χώρας μας και τις αξίες που θα προέκυπταν. Σήμερα όμως βλέπουμε μια ανησυχητική τάση, κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να προασπίσει το Ευρωκοινοβούλιο τα δημοκρατικά μου δικαιώματα σαν βουλευτό. Η κυρία Βάρτορα. Κύριος, με συγχωρείτε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σε προηγούμενη παρέμβαση αναφέρθηκα σε ένα πρόβλημα που έχει διαπιστωθεί από πολλές μελέτες Αναφέρομαι στην αποδυνάμιση της δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παγκόσμια. Έχουμε λοιπόν ένα δίκτυο που αναφέρεται στην ελευθερωρία των ΜΜΕ. Αυτό αφορά ειδικότερα τα νέα κράτη-μέλη. Σας δίνω λοιπόν το παράδειγμα της Σλοβενίας. Στον κατάλογο της ελευθερίας των ΜΜΕ η Σλοβενία είναι 7 θέσεις χαμηλότερα από ό,τι πριν στις μεταβατικές χώρες μπορούμε να δούμε πολύ ευάλωτη κατάσταση διότι τα μέσα, τα ΜΜΕ είναι κάτω από την επιρροή του κεφαλαίου η κοινωνική κατάσταση είναι άσχημη και δεν υπάρχει και επαγγελματική πείρα. Υπάρχει συνεπώς μια γενική τάση, αλλά θα έπρεπε να υπογραμμίσουμε την ύπαρξή της και ζητώ από τα κράτη-μέλη και την Κομισιόν να αναπτύξουν μια στρατηγική αποτελεσματική για την καταπολέμηση της έλλειψης ελευθερίας για το ΜΜΕ. Πρέπει να είμαστε αντικειμενικά ενημερωμένοι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Το Μάρτιο φέτος το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε από την Κούβα να αφήσει ελεύθερους τους πολιτικούς κρατούμενους. Ε, αιτία ήταν ο τραγικός θάνατος αυτούς λόγω απεργίας πείνας. Όμως ε, το κουβανικό καθεστώς αντέδρασε κοινικά και με βάση αυτά τα δεδομένα είναι εκπληκτικό ότι η Ισπανική Προεδρία απαιτεί να αλλάξει στάση η Ευρωπαϊκή Ένωση και να απομακρυνθούμε από τη σκληρή γραμμή έναντι της Κούβας. Τα τελευταία χρόνια άναξαν πολλά, αλλά εξακολουθεί να είναι δικτατορία η Κούβα. Εγώ θεωρώ πως μπορεί να υπάρξει προσέγγιση με την Κούβα μόνο όταν είναι διατεθειμένο να κάνει μια χειρονομία το κομμουνιστικό καθεστώς. Δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων από πλευράς εξωτερικής πολιτικής. Πρέπει να είμαστε συνεπείς και αξιόπιστοι. Ο κύριος Ντόιτς. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, χιλιάδες Ευρωπαίοι περιμένουν τη βοήθειά μας λόγω των πλημμυρών. Είναι οι Ευρωπαίοι της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης χιλιάδες άνθρωποι, εκατομμύρια άνθρωποι περιμένουν τη βοήθειά μας. Τσέχοι, Πολωνοί, Σλοβάκοι, Ούγγροι, εκατομμύρια άτομα είναι θύματα των πλημμυρών αυτών που κρατούν βδομάδες, πολλές βδομάδες με τεράστιο ρυθμό θυμάτων. Στα Ουγγαρέζικα λέμε όταν δίνουμε γρήγορα δίνουμε δύο φορές. Τρεις φορές θα δώσουμε αν δώσουμε πολύ γρήγορα και αυτό κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό πρέπει να κάνει και το Κοινοβούλιο. Αλλά δεν πρέπει να βιαστούμε και πάρα πολύ, πρέπει να σκεφτούμε λίγο τι θα πάρουμε, αλλά ταυτόχρονα να προσφέρουμε βοήθεια γρήγορα. Και αυτό ζητάμε και από την ε, Κομισιόν. Πρώτες, κάποιες αναγγελίες. Πρώτον, μπλε κάρτες δεν υπάρχουν. Δεύτερον, αναφέρω τα ονόματα όπως υπάρχουν στον κατάλογο μπροστά μου. Η κυρία Γκουτιέρης Κοτίνα, επόμενη. Κοτίνα, συγγνώμη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μιλώ υπέρ των μαθητών των Ευρωπαϊκών Σχολείων, των οποίων τα προσόντα δεν αναγνωρίζει το Ισπανικό Υπουργείο Παιδείας. Είναι όλοι σχεδόν παιδιά υπαλλήλων ε, της Ένωσης και αντιμετωπίζονται με άδικο τρόπο. Η έλλειψη ε, που επέβαλε πρόσφατα το Υπουργείο μειώνει κατά μισό ή ένα ποντό τους φοιτητές που σπούδασαν στα ευρωπαϊκά σχολεία, που μιλούν πολλές καινές γλώσσες και που σημαίνει ότι τώρα όταν θέλουν να μπουν σε σταδιοδρομίες που απαιτούν υψηλό ποσοστό ε, ε, βαθμών μένουν πίσω. Αυτό είναι παράνομο διότι η Ισπανία έχει υπογράψει μια σειρά συμφωνιών που δεν τηρεί και δεύτερον διότι αποτελεί βασική διάκριση. Δεν μπορεί να θεωρούμε ότι είμαστε ευρωπαϊκή χώρα όταν αντιμετωπίζουμε με διακριτικό και άδικο τρόπο τους, φοιτητές, τους μαθητές των σχολείων Σας Ευχαριστώ. Ο κύριος Μέλλο. Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να, να καταγγείλω ένα έγκλημα κατά του περιβάλλοντος. Τα τέλειωτα άχρηστα απορρίμματα, πολύ επικίνδυνο, απορρίφθηκαν σε μία ε, περιφέρεια στο, στη Βόρεια Πορτογαλία. Ε, μολύνθηκε το έδαφος, μολύνθηκαν τα ύδατα. Πρόκειται για ψευδάριο, αρσενικό, και οι αρχές της Πορτογαλίας, αν και ενημερώθηκαν, δεν παρενέβησαν σε αυτή, με την κυβέρνηση τη σοσιαλιστική τώρα. Ε, έχουμε λάβει μια απάντηση σε, σε ερώτηση βουλευτού λέγοντας ότι είχε εξασφαλιστεί μια παρέμβαση κατάλληλη. Θα ήθελα λοιπόν να παρέμβουν όμως και ε, τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχω ήδη αναφερθεί στην Κομισιόν και κάνω έκκληση σήμερα στο Ευρωκοινοβουλίο και ελπίζω ότι θα υπάρξει ένα ψήφισμα που θα υπερψηφιστεί. Ο κύριος ευχαριστώ επιτέλους πρόεδρε. Ε, επιτυγχάνεται η ισότητα ανδρών γυναικών. ευαναβαίνει στα 65 ε, το όριο συνταξιοδότησης. Ε, παλιά αυτό είχε προβλεφθεί με βαθμίο τρόπο που θα ε, επέτρεπε στην Ιταλία μόνο το 2018 να υπάρξει η εξίσωση. Ωστόσο η κυβέρνηση αμέσως προσαρμόστηκε και χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν ήταν δικαιολογημένη και αιτιολογημένη η απόφαση. Η αποταμίευση που θα η εξοικονόμηση που θα προκύψει πρέπει να εξασφαλίζεται Πρέπει να εξασφαλίζει, η οθόνη ε, μέτρα αντισταθμιστικά για να, για να υποστηριχθεί ακριβώ η εργασία των γυναικών. Προηγουμένω ε, μίλησε η κυρία Αλφάνο για το νόμο για τι υποκλοπές. Αντίθετα, ωστόσο, από αυτό που είπε, δεν είναι νόμο. Ο νόμος ε, θα επιτρέψει την εξισορρόπηση του δικαιώματο στην προσωπική ζωή και του δικαιώματο στην ενημέρωση. Και όλα αυτά τα λαμβάνει υπόψη το τελικό κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η κυρία Ζαμπρόσκα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λούτζα ο Λούτζι Ραπετζάντα, επίσκοπος στην Τουρκία, δολοφονήθηκε και θα ήθελα να κάνω δύο σχόλια. Πρόκειται βεβαίω για ψυχική αστάθεια λέει, του δολοφόνου, αλλά αυτό το επιχείρημα, το επιχείρημα το χρησιμοποιούν πολύ συχνά για δολοφονίες στην Τουρκία πρωτοί καν ξεκινήσει η ανάκριση. Είναι πολύ βολικό κάτι τέτοιο να, ε, να αποκαλούμε ε, εξτρεμιστή, ε, φανατικό το δολοφόνο. Κανένας από τους Ευρωπαίους πολιτικούς δεν αντέδρασε για αυτή την δολοφονία και αυτό είναι αποτέλεσμα των μίντια εάν πρόκειται για καθολικό επίσκοπο υπάρχουν διάφορες αντιδράσεις. Υπάρχει μίσος ή καμπάνια ενεργοποίησης. Θα ήθελα λοιπόν τα θεσμικά όργανα της Ευρώπης να παρακολουθήσουν πολύ προσεκτικά αυτή τη δολοφονία και να ασχοληθούν με τη δίωξη των χριστιανών στις ε, διαπραγματεύσεις ένταξης της Τουρκίας. Ο κύριος Higgins τελευταίος. Κυρία Πρόεδρε, απόψε άντρες, γυναίκες και παιδιά από τρεις κοινότητες του Δουβλίνου στην εσωτερική, στο εσωτερικό της πόλης διαμαρτυρήθηκαν στο Δημαρχείο για να μην κλείσει η πισίνα τους, η δημοτική. Το Δημοτικό Συμβουλίο λέει ότι δεν έχει λεφτά πια. Σε αυτές τις κοινότητες που έχουν φυγεί από υψηλή ανεργία, το να κλείσει κανεί τις πισίνες αυτές είναι βανταλισμός κοινωνικός. Το κλείσιμο σημαίνει μεγάλες περικοπές από την κυβέρνηση ε, που υποστηρίζει άλλωστε και η Κομισιό. Το κόστος λειτουργίας αυτών των πισινών ε, θα ήταν ένα εκατομμύριο ευρώ. Εν τω μεταξύ 30 δις ευρώ ε, ρίχνει η κυβέρνηση για να δημιουργήσει νέα κεφαλαία για τις τράπεζες, για να διαρθρώσει τα κεφαλαία τους.